διαπραγματεύσεις. Τώρα περνάμε στην ημερήσια διάταξη μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης. Δίνω το λόγο στην εισηγήτρια κυρία Γκαρντίνη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σήμερα νομίζω ότι θα γράψουμε μία πολύ ωραία σελίδα της ευρωπαϊκής ιστορίας και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ε, τους εμπλεκόμενους, αρχίζοντας από τους εισηγητές όδης, αλλά και ολόκληρο το κοινοβούλιο, το οποίο με την ευελιξία του και την δυνατότητα να ε, διαβλέψει την ενίσχυση αυτού του μηχανισμού πολιτικής, πολιτικής προστασίας, να κατάφερε να μπορέσει να ξεπεράσει ορισμένες αμφιβολίες κρατών μελών, έτσι ώστε η πολιτική προστασία να μην θεωρηθεί παρεμβατισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωβαρόμετρο δείχνει ότι οι πολίτες θέλουν την πολιτική προστασία και θέλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλάι τους τη στιγμή που οι τοπικές και περιφερειακές αρχές δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν έκτακτες καταστάσεις. Είδαμε τι ε, έγινε με τις πυρκαγιές του καλοκαιριού στην Πορτογαλία και την Ελλάδα, όπου χάθηκαν πολλές ε, ζωές πέρα από τις ε, οικονομικές ζημίες. Γι' αυτό χρειάζεται αυτός ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, γιατί δεν μπορεί να γίνει αντιμετώπιση σε τοπικό ή κρατικό επίπεδο πάντα. Ένα χρόνο μετά την ανακοίνωση της Επιτροπής και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για τη σπουδή με την οποία ε, αντιμετώπισε το θέμα ο Επίτροπος Στυλιανίδης, έχουμε το RESC-EU. Το RESC-EU είναι ένα νέο μέσον που απαρτίζεται από επιπρόσθετους πόρους σε σχέση με τους προϋπάρχοντες και που είναι των κρατών μελών. Γιατί το RESC EU θέλει ακριβώς να μπορέσει να ανταποκριθεί άμεσα εκεί όπου χρειάζεται, μέσα στα πλαίσια και της πρόληψης και της προετοιμασίας έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις φυσικές καταστροφές είτε όταν πρόκειται για ατυχήματα τα οποία προκύπτουν από την χρήση χημικών ουσιών, πυρηνικά ατυχήματα και ούτω καθεξής. Υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι οι πυρκαγιές είναι υπεύθυνες για το 20% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε αυτόν τον ενισχυμένο μηχανισμό. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ως Ιταλίδα να σας υπενθυμίζω τον Τζουζέπε Τζαμπερλέτη που είναι ο θεματοφύλακας της πολιτικής προστασίας και θα ήθελα να του αφιερώσω αυτή την ημέρα και αυτή την εργασία κύριε Επίτροπε γιατί πέρα από ένα είδος εράσμου το οποίο θεσμοθετήθηκε και που αποτελεί ε, έναν κοινό παρονομαστή όλων, υπάρχει και ο μηχανισμός αναγνώρισης για εκείνους ε, οι οποίοι διακρίθηκαν στο τομέα της πολιτικής προστασίας. Γι' αυτό θα ήθελα να ε, θυμίσω την ύπαρξη αυτού του μεγάλου ανθρώπου και νομίζω ότι σήμερα μας στέλνει και εκείνος ένα μεγάλο χαμόγελο για αυτή την εργασία. Ευχαριστώ κυρία Γκαρντίνη. Ναι, και εγώ θα ήθελα να πω ότι γνωρίσαμε πολύ καλά τον κύριο Τζαμπερλέτη, ο κύριο Ζόφκο από την Επιτροπή, η κυρία Ζόφκο, από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να κάνω κάποια σχόλια, να συγχαρώ την κυρία Γκαρντίνη, διότι έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά στο θέμα της έκθεσής μας, την πολιτική προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον Επίτροπο κύριο Στυγιανίδη. Ήμουν εισηγήτρια προς γνωμοδότηση από την Επιτροπή Ανάπτυξης και θέλαμε να τονίσουμε την ανάγκη να, ενισχυθεί, να ενισχυθούν και οι εθνικές ικανότητες πολιτικής προστασίας και οι διεθνείς συνεργασίες, επιτρέποντας τους μηχανισμούς στις διάφορες χώρες ε, μέλη να λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους. Το νέο εργαλείο πρέπει να έχει στόχο την πρόληψη κινδύνων. Είχαμε πολλές πυρκαγιές ε, δασών τα τελευταία χρόνια, ιδίως στην Νότια Ευρώπη και χρειάζεται από πλευράς μας να υπάρξει μια ισχυρή αντίδραση. Θα ήθελα να ζητήσω οι χώρες εκείνες που δεν μπορούν να μετάσχουν πλήρως, να λάβουν κάποια χρηματοδότηση για τη μεταφορά, 50% ενδεχομένως. Αυτό για την Κροατία, για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντικό. Η Κροατία χρειάζεται μια σειρά υποστηρικτικών δράσεων για όλα τα μέτρα ε, πολιτικής προστασίας. Επίσης, ο μηχανισμός Rescue θα πρέπει να επιτρέπει πάντα στα κράτη-μέλη να ελέγχουν την ανάπτυξη των δυνάμεων στο κράτος, στα κράτη-μέλη. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν για τον μηχανισμό αυτό που θα επιτρέψει στους πολίτες της Ένωσης να μην αισθάνονται απομονωμένοι πλέον. Ευχαριστώ. Ο κύριο Στυλιανίδη, ο επίτροπο, έχει το λόγο και εγώ τον ευχαριστώ για την παρουσία του στην Ολομέλεια σήμερα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, μίλησα στη, στο Κοινοβούλιο πριν από ένα χρόνο περίπου, παρουσιάζοντας την πρότασή μας για την ενίσχυση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα, μετά από ένα χρόνο, το Κοινοβούλιο ψηφίζει την πλέον φιλόδοξη, το πλέον φιλόδοξο σύστημα πολιτικής προστασίας στην Ευρώπη που έχει υπάρξει ποτέ. Σήμερα το Κοινοβούλιο ψηφίζει κάτι που ήταν πολιτικά διανόητο πριν από λίγα χρόνια. Είμαστε φίλοι εδώ τώρα και θα σας τα πω με ειλικρίνεια. Ήταν πολύ απαιτητική δουλειά, πολύ δύσκολη δουλειά να πείσω τα κράτη να δεχθούν αυτή την προσέγγιση. Εν τέλει όμως καταφέραμε και υλοποιήσαμε αυτόν τον πολύ φιλόδοξο κοινό στόχο. Σήμερα λοιπόν είμαι πραγματικά περήφανος που είμαι Ευρωπαίος. Θέλω Πρώτα πρώτα να, να ευχαριστήσω ειλικρινά την εισηγήτρια κυρία Γκαρντίνη για την ηγετική θέση που έλαβε στην, στο να προωθήσει το σημείο αυτό στο Κοινοβούλιο και όλους τους συναδέλφους την κυρία Ζόφκο τον κύριο Ενάντες και όλους τους σκιώδεις εισηγητές από τις πολιτικές ομάδες τις πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου, το Κοινοβούλιο ολόκληρο που υποστήριξαν με πάθος αυτό το ρηξικέλευθο μέτρο. Συνάδελφοι, με την πολιτική σας υποστήριξη το Rescue θα είναι εκεί παρόν στις επόμενες δασοπυρκαγιές. Και χάρη στην δική σας αφοσίωση στον κοινό μας στόχο, για την προστασία των πολιτών μας, για την διάσωση ανθρώπινων ζωών και των σπιτιών τους. Πραγματικά ζητήσατε εγγυήσεις για καλύτερη και άμεση διαθεσιμότητα ανταπόκρισης στις καταστροφές. Και σήμερα μπορώ να σας πω το εξής. Συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη-μέλη για να ξεκινήσουμε το συντομότερο δυνατό την μεταβατική φάση του rescue, όπως το λέμε, ούτως ώστε να μπορούν να υπάρξουν ικανότητες ε, ανταπόκρισης της κρίσης για την Ευρώπη ήδη φέτος. Η ενημέρωση και οι πληροφορίε που παίρνω από τα κράτη-μέλη μέχρι τώρα είναι πολύ θετικέ και ευχαριστώ και εγώ τα κράτη-μέλη σήμερα για την θετική τους προσέγγιση. Βέβαια, μην βαφκαριζόμαστε. Δεν θα σταματήσουν οι φυσικέ καταστροφέ. Αντίθετα, θα γίνονται συχνότερε και πιο έντονε λόγω τη αλλαγή του κλίματο. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το νέο αυτό φαινόμενο της αλλαγής του κλίματος όσο καλύτερα μπορούμε. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε με το Rescue είναι να εξοπλίσουμε καλύτερα και τους εαυτούς μας και τα κρατημέλη για να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις καταστροφές από την αλλαγή του κλίματος. Η νέα αυτή νομοθεσία κυρίε και κύριοι δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη και την προπαρασκευή. Το Κοινοβούλιο κατέστησε σαφές ότι τούτο ήταν προτεραιότητα για εσά και κάναμε ό,τι μπορούμε για να θεσπίσουμε ένα σύστημα που παρέχει περισσότερη υποστήριξη στα κράτη για την ανταλλαγή πληροφοριών και για να διδαχθεί το ένα από το άλλο. Συνάδελφοι, σήμερα με μετριοφροσύνη μπορώ να πω ότι από... χαράσουμε το ξεκίνημα μιας νέας εποχής πολιτικής προστασίας στην Ευρώπη. Μιλάμε για μια Ευρώπη που προστατεύει. Αυτό το οφείλουμε, όπως είπα, στους πολίτες μας. Κλείνω επαναλαμβάνοντας ότι θα πρέπει όλοι να είμαστε περήφανοι λόγω του επιτεύγματος αυτού και θέλω εκ νέου να σας ευχαριστήσω για την αφοσίωση και την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την Επιτροπή Προϋπολογισμών ο κύριος Φερνάντες ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρώπη που προστατεύει αποτελεί μία αναγκαιότητα. Η προστασία της ανθρώπινας ζωής θα πρέπει να είναι το βασικό μας μέλημα. Το 2017 στην Πορτογαλία ζήσαμε μία μεγάλη τραγωδία. Πάνω από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Αυτό δεν μπορεί να επαναληφθεί. Ο νέος αυτός μηχανισμός δείχνει την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βλέπουμε ότι αυτό που έχει σημασία είναι ο επιμερισμός των ευθυνών, ιδιαίτερα όσον αφορά την πολιτική προστασία. Και αυτό δείχνει ακριβώς ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να στοιχηματίζουμε στην πολιτική προστασία και η προστασία είναι το βασικό μας μέλημα. Επίσης, πολλοί υπουργοί οικονομικών δεν δέχτηκαν αυτή τη συμφωνία και τι έκαναν, διαπραγματευτήκαν ένα ποσό 100.000 ευρώ, δηλαδή ένα μελιτέο ποσό για το 2019. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την δέσμευση του κυρίου Στυλιανίδη και της κυρίας Γκαρντίνη, έτσι ώστε να φτάσουμε σε μία συμφωνία που δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση σώζει ζωές και αυτό πραγματικά αξίζει. Η κυρία Μίλναρ δεν είναι παρούσα, άρα περνάμε στις πολιτικές ομάδες. Για το ΕΛΚ ο κύριος Γκαμπής για 1,5 λεπτό. Θα ήθελα όλοι να τηρείτε το χρόνο σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η Ευρώπη δημιουργείται μέσω της αλληλεγγύης και της αδελφοσύνης μεταξύ των λαών της. Αυτή είναι μια αρχή που σήμερα περισσότερο παρά πρέπει να υπενθυμίσουμε εδώ στο ημικύκλο στο Τρασβούργο. Η αλληλεγγύη μεταξύ των Ευρωπαίων δημιουργείται από κάτω προς τα πάνω και με βάση αυτή την πιο βασική ανάγκη που είναι η αντιμετώπιση των απροβλέπτων ε, θεομηνίων όπως είδαμε στις τεράστιες πυρκαγιές στην ε, Πορτογαλία και την Γαλλική του 2017. Όμως πρέπει να είμαστε και έντιμοι μεταξύ μας. Κάτι λείπει όταν η Ευρώπη δεν είναι η πρώτη που να ανταποκρίνεται όταν υπάρχει μια τέτοια θεομηνία. Γι' αυτό θεωρώ ότι η δημιουργία του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας είναι ένα καλό εργαλείο που μπορεί να συνδυαστεί με την πρόταση για αυτό το σώμα Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης. Και έτσι θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να είμαστε περήφανοι για την Ένωση, για να δείξουμε ότι μέσω της ενότητας μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις προκλήσεις που έχουμε ενώπιόν μας. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, τη συνάδελφο Γκαρντίνη, για την εργασία της για το θέμα αυτό, για το καλό αποτέλεσμα που επέτυχε και για τη λειτουργικότητα και την άμεση επίπτωση που θα έχει αυτός ο μηχανισμός στο μέλλον στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε. Για τους σοσιαλιστές, ο κύριος Ανδρουλάκης. Ε, παρακαλώ, Νίκο, δυόμιση λεπτά. Τελευταία χρόνια, σε πολλούς από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι θεσμοί μοιάζουν απόμακροι, ακόμα και εχθρικοί όμως στην περίπτωσή μας η αγωνία τους για καλύτερη προστασία από φυσικές καταστροφές αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη στην προσπάθειά μας να καταστήσουμε τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας ένα πραγματικό εργαλείο αλληλεγγύης δημιουργώντας το resceu. σήμερα η ανθρωπιά και η στήριξη των λιγότερο δυνατών και η περιβαλλοντολογική ηθική είναι νικητές. η αφορμή για τη συγκεκριμένη πρόταση ήταν οι καταστροφικές πυρκαγιές στην πορτογαλία. κανείς όμως δεν μπορούσε να φανταστεί ότι λίγο πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις μια νέα τραγωδία θα έπληκε την ευρώπη. αυτή τη φορά στο μάτι λίγο έξω από την αθήνα με πάνω από 100 νεκρούς. αυτά τα γεγονότα κατέστησαν σαφές σε όλους ότι πρέπει να προσφέρουμε μια ουσιαστική απάντηση στις ανησυχίες των πολιτών. Σε αυξανόμενε φυσικές καταστροφές, λόγω κλιματικής αλλαγής ή ανεπαρκή προετοιμασία από τις εθνικές αρχές, δεν μένουμε παρατηρητές, αλλά δίνουμε μια ισχυρή απάντηση. όλοι μαζί με περισσότερη οργάνωση μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα από ό,τι ο καθένας μόνος του. ο δρόμος τη πολιτική ενοποίηση είναι μακρύ και γεμάτος εμπόδια που βάζουν οι θειασότες μιας Ευρώπης, όπου η αλληλεγγύη δεν είναι αυτό αλλά μέσο με κόστο που δεν θέλουν να αναλάβουν ο ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτική προστασία αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έμπρακτη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. δημιουργούμε το resceu μια ευρωπαϊκή δεξαμενή μέσων όπω πυροσβεστικά ελικόπτερα και αεροπλάνα τα οποία θα αγοραστούν με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το 80 90% των συνολικών εξόδων διασφαλίζοντας ότι καμία χώρα δεν θα μείνει ξανά αβοήθητη. παράλληλα για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης έως 75% για τη συντήρηση των εθνικών μέσων. η βοήθεια αυτή σε χώρες όπως η ελλάδα που η αδυναμία επισκευής λόγω της οικονομικής κρίσης έχει περιορίσει πάρα πολύ τη δράση των εθνικών μέσων είναι απαραίτητη. τέλος ενισχύουμε την πρόληψη διατηρώντας ανώθευτα τα χαρακτηριστικά της αλληλεγγύης. απορρίψαμε την πρόταση του συμβουλίου που προέβλεπε την εισαγωγή ποινών για τι χώρε που ζητούν συχνά την ενεργοποίηση του μηχανισμού. αντιθέτω δίνουμε τη δύναμη στην επιτροπή να εξετάσει τα μέτρα πρόληψη του συγκεκριμένου κράτου και όπου χρειάζεται να παρεμβαίνει να υπάρχουν συστάσει για βελτίωση ή ενίσχυση των εθνικών σχεδίων προστασία. όλοι οι ευρωπαίοι πολίτε ανεξάρτητα του κράτου μέλου που κατοικούν πρέπει να νιώθουν ασφαλεί και να ξέρουν ότι η ένωση μπορεί να του βοηθήσει με πρακτικό και αποτελεσματικό τρόπο σε περίπτωση μια έκτακτης ανάγκης. Για την, του συντηρητικούς ο κύριος Γκέρικε. 1,5 λεπτό παρακαλώ. Από πλευρά ε, των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών θέλω να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Γκαρντίνη η οποία ασχολήθηκε με αυτή τη διοργανική συμφωνία που ανταποκρίνεται σε όλα τα ε, αιτήματά μας και συνεργάστηκε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τι άλλε πολιτικέ ομάδε. Έτσι θα έχουμε ιδιαίτερε υπηρεσίε διάσωση που θα βοηθούν τα κράτη-μέλη αν έχουν συμπεραστεί από τα γεγονότα οι δικέ του υπηρεσίε. Όπω ιδιαίτερα κατά τι ε, δάσοπυρκαγιέ ε, τον περασμένο καλοκαίρι. Ελπίζουμε μέχρι το καλοκαίρι να έχουμε ειδικά πυροσβεστικά αεροπλάνα για να καταπολεμήσουμε τι πυρκαγιέ που κατά πάσα πιθανότητα και πάλι θα προκύψουν. Θεωρώ ότι πετύχαμε λοιπόν τη συνεργασία Κάτι που σπάνια έχουμε επιτύχει στο μέλλον, ούτως ώστε η αντιμετώπιση των καταστροφών να βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές. Και έτσι νομίζω ότι είμαστε πρωτοπόροι όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά παγκοσμίως. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Γιάτενμα και 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ και την κυρία Γκαρντίνη Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι τελικά η κύρια ευθύνη για την πολιτική προστασία εξακολουθεί να παραμένει στα χέρια των κρατών μελών. Οι ενωσιακοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν μόνο ως ίστατη προσφυγή. Κανένα κράτος μέλος ούτως ή άλλως όμως δεν θα πρέπει να δώσει ως υπεργολαβία την πολιτική προστασία σε άλλες χώρες. Αυτό θα ήταν και επικίνδυνο και ανεύθυνο. Ξέρουμε ότι όταν ε, υπάρχει μια θεομηνία πρέπει κανείς να δράσει ε, τάχιστα. Διότι τα πρώτα λεπτά, οι πρώτες ώρες ε, είναι πιο σημαντικές για την αντιμετώπιση της. Αν περιμένουμε να έρθουν από αλλού οι αρμόδιοι της πολιτικής προστασίας για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, τότε οι επιπτώσεις θα είναι πραγματικά τραγικές. Η πρόληψη φυσικά είναι πάντα καλύτερη από την αντιμετώπιση, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ έχει ρόλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να στηρίξει τα κράτη-μέλη και για την ε, πρόληψη και για την αντίδραση βεβαίω. Όλα αυτά πρέπει να βελτιωθούν και βεβαίω και η διαλειτουργικότητα ε, του εξοπλισμού είναι αναγκαία. Αλλά το κάθε κράτος μέλος θα πρέπει αυτό και μόνο να έχει την ε, αρμοδιότητα για να έχει διαθέσιμο το κατάλληλο εξοπλισμό εάν υπάρξει πρόβλημα αλλά και η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών είναι βεβαίως και αυτή πολύ σημαντική. Αναφέρθηκαν οι δασοπυρκαγιέ. Και εδώ η πρόληψη είναι ιδιαίτερα σημαντική για να αποφεύγονται. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Παπαδημούλης για την ΚΟΕ, ένα λεπτό. Είναι μία από τις λίγες θετικές ειδήσει που παράγουμε ως ευρωπαϊκή θεσμή το τελευταίο διάστημα και αυτό το οφείλουμε στην πίεση του ευρωκοινοβουλίου στις θετικές προσπάθειες του επιτρόπου στυλιανίδη και στη συνεργασία ευρωκοινοβουλίου Κομισιών που έκαμψαν τις αντιρρήσεις ορισμένων κρατών μελών. Γιατί ήρθαν και τα γεγονότα να βοηθήσουν. Τα τραγικά γεγονότα. Οι μεγάλες πυρκαγιές στην Πορτογαλία. Φωνικές οι πυρκαγιές στην πατρίδα μου την Ελλάδα και οι πλημμύρες φωνικές, οι σεισμοί στην Ιταλία, με νεκρούς επίσης, αλλά και οι μεγάλες πυρκαγιές στη Σουηδία που έκαναν και τους βόρειους τα βόρεια κράτη-μέλη να καταλάβουν ότι η κλιματική αλλαγή δεν απειλεί μόνο τον Νότο και ότι χρειαζόμαστε μια επικουρική δύναμη ευρωπαϊκή να ενισχύει τις προσπάθειες των κρατών μελών. Και έπαψε αυτή η ευρωτσιγκουνιά. Και έχουμε περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη. Και η τελική πρόταση είναι βελτιωμένη χάρη στην επιμονή του Ευρωκοινοβουλίου και κινείται σε θετική κατεύθυνση. Και γι' αυτό νομίζω ότι έχει και μια ευρύτερη στήριξη μες στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ακούσαμε τις απόψεις των πολιτικών ομάδων. Κάποιοι αγορητές ή, ατομικά. Ο κύριος Μάντελ, 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι. Ο χειμώνας στην Αυστρία απέδειξε ότι οι υπηρεσίες διάσωσης, οι εθελοντές, οι πυροσβέστες και οι άλλες ε, δυνάμεις για την αντιμετώπιση είναι θαυμάσιες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Εμείς είμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να έχουμε την ε, ε, δυνατότητα να μην χρειαζόμαστε βοήθεια εκ των έξω όταν προκύψουν απρόβλητες καταστροφές οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν σε διαπεριφερειακό επίπεδο. Είναι σωστό λοιπόν που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα μηχανισμό αντιμετώπισης καταστροφών. Και συμμερίζουμε αυτό που είπαν ήδη ε, επανειλημμένα οι συνάδελφοι, ότι εμεί, ω Κοινοβούλιο βελτιώσαμε ιδιαίτερα την έκθεση. Είναι λιγότερο συγκεντρωτική, λιγότερο γραφειοκρατική και χαίρομαι που η Προεδρία του Συμβουλίου είναι τώρα στην ε, Αυστρία και αυτή θα ολοκληρώσει αυτή την επιτυχία. Και εμείς επίσης μπορούμε να κρίνουμε το τελικό αποτέλεσμα. Διότι η αρχική πρόταση της Κομισιόν που προέβλεπε κέντρα ε, ελέγχου και παροχής εντολών, καταλήγουμε τώρα σε ένα πακέτο που στηρίζει περισσότερο την συνεργασία και πρώτα απ' όλα την ενίσχυση των περιφερειακών και τοπικών μηχανισμών ασφαλείας. Αυτό είναι το παράδειγμα της Αυστρίας και έπαιξε ένα ρόλο νομίζω στη διαμόρφωση της τελικής πρότασης. Και βεβαίως θα πρέπει κυρίως να βασιζόμαστε στις ε, δικές μας δυνάμεις. Ο κύριος Ζωρίνιο, Κάρλος, παρακαλώ λεπτό. Σήμερα κάναμε ένα σημαντικό βήμα για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας έτσι ώστε να μπορέσουμε συντονισμένα να συνδράμουμε τα κράτη-μέλη. Οι καταστροφές ήταν συντριπτικές για ολόκληρη την Ευρώπη, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Γι' αυτό χρειάζεται αυτός ο πολιτισμός πολιτικής προστασίας παντού και όχι μόνο στο Νότο και γι' αυτό χρειάζεται και η κατάλληλη πόλη. Πιστεύω ότι η δημιουργία αυτού του αποθεματικού ΡΕΣΚΙΓΙΟΥ είναι ύψη τη σημασίας και η συζήτηση και η έκθεση μας επέτρεψαν να ολοκληρώσουμε αυτή την προσπάθεια, να συγχαρούμε την εισηγήτρια και ελπίζουμε να έχουμε και την στήριξη των κρατών μελών για να μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε όλους τους κινδύνους. Ε, κύριε Επίτροπε, όμως αυτή η πολιτική ε, δεν μπορεί να αναβληθεί για το μέλλον. Θα πρέπει να υπερβούμε τους γραφειοκρατικούς ε, μηχανισμούς και αυτό μέσα στα πλαίσια και του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου 21-27. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το χρονοδιάγραμμα της πρότασης νομοθετικού περιεχομένου. Εάν λοιπόν δημοσιευτεί σήμερα, ήδη θα ήταν αργά. Θα πρέπει να αποτρέψουμε τις φυσικές καταστροφές. Χρειάζονται οι πολίτες το ήδη. Φερέιρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία των κρατών μελών, ιδιαίτερα για τις καταστροφές μεγάλων διαστάσεων. Χρειάζεται συντονισμός προσπαθειών και επιμερισμός ευθυνών. Η Ευρώπη δεν έχει κάνει ό,τι μπορούσε σε αυτό το τομέα. Η κατάσταση το 2017 στην Πορτογαλία ε, καταδεικνύει την κατάσταση. Οι πυρκαγιές στην ε, Πορτογαλία ήταν καταστροφικές και δυστυχώς θα υπάρξουν και περικοπές από όσο προβλέπεται, ακόμα και για την πρόληψη των καταστροφών. Δυστυχώς οι καταστροφές πλήττουν χώρες που δεν έχουν τόσο σοβαρά μέσα στη διάθεσή τους για να τις αντιμετωπίσουν. Θα πρέπει λοιπόν να τονίσουμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν την εποπτεία αυτού του μηχανισμού. Διαφορετικά, αν υπάρχει αποκέντρωση, τότε ελοχεύουν κίνδυνοι και πιστεύω ότι δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους σε εθνικό επίπεδο. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Ε, Ρουίθ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που αρχίζει να λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός που σημαίνει περισσότερη Ευρώπη, Ευρώπη αλληλεγγύης, ούτω ώστε να προλαμβάνουμε και να αντιμετωπίζουμε και να απαλύνουμε τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών. Αλλά τονίζω ότι πρέπει να τροποποιηθεί το Ταμείο Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύης που πρέπει να δώσει αποζημιώσεις για τις φυσικές καταστροφές. Είναι σημαντικό, όπως έχουμε ζητήσει, να συμπεριληφθεί και το περιβάλλον να ληφθεί η υπόψη η οικονομική ζημία από τις περιβαλλοντικές καταστροφές για να δίδονται αποζημιώσεις. Είναι σημαντικό οι περιφέρειες που θα μπορέσουν να υποφεληθούν από αυτό το ε, ταμείο να υπολογίζονται με βάση το τοπικό ΑΕΠ και όχι το ΑΕΠ ολόκληρη τη αλληλεγγύη. Έτσι μόνο θα αντιμετωπίσουμε τι ε, ε, καταστροφέ που αντιμετωπίζουν διάφορε περιοχέ που έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Θέλω λοιπόν να κάνω μία έκκληση να βοηθήσει και αυτό το Ταμείο Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μεταρρύθμιση του κανονισμού του. Και σας εύχομαι κάθε επιτυχία κύριε Επίτροπε. Ο κύριο Μαρια, ένα λεπτό. Οι φυσικές καταστροφές δυστυχώς είναι στην ημερήσια διάταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω φυσικά των κλιματικών αλλαγών. Και είχαμε τεράστιες καταστροφές, είχαμε τις ε, φωνικέ πλημμύρε στη μάντρα τη Αττικής, τι φωνικέ πυρκαγιέ στο Μάτι με 100 νεκρούς, πυρκαγιές επίσης φωνικές στην Πορτογαλία, σεισμούς με νεκρούς στην ε, Ιταλία. Όλα αυτά δείχνουν ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέτει ένα μηχανισμό πολιτικής προστασίας αποφασιστικό που να ενσωματώνει στην πράξη την αρχή της αλληλεγγύης. Και νομίζω ότι τα βήματα που γίνονται είναι σε μια θετική κατεύθυνση. Θα πρέπει να καταλάβουν τα κράτη-μέλη ότι δεν μπορούν να επιβάλλουν ποινές στις χώρες οι οποίες θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν αυτό το μηχανισμό διότι η αξιοποίηση αυτού του μηχανισμού προέρχεται δυστυχώς λόγω των φυσικών καταστροφών. θεωρώ ότι πρέπει να πάρουμε ακόμη πιο αποφασιστικά μέτρα να στηρίξουμε τις χώρες που υφίστανται τις φυσικές καταστροφές και αυτές κυρίως είναι οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου. ευχαριστώ. Η κυρία ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή συζήτηση καταδεικνύει άλλη μια φορά σαφέστατα ότι η προστασία από τις καταστροφές και αντιμετώπιση αφορά πολλά θέματα, τη χωροταξία, την προστασία του περιβάλλοντος, την κατάρτιση, πρώτα απ' όλα βεβαίως η πρόληψη. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τέτοιες καταστροφές. Χρειαζόμαστε καλή παρακολούθηση και νομίζω ότι η συζήτηση και η απόφαση που ελπίζω ότι θα ληφθεί για αυτό το μηχανισμό θα συμβάλλει ιδιαίτερα ούτως ώστε στο μέλλον να μπορούμε να πούμε στους ε, συμπολίτες μας ότι αν υπάρξουν θεομηνίες η Ευρώπη βοηθάει όλοι μαζί. Δεν αφήνουμε μόνο τους, ε, τα κράτη-μέλη, τις περιφέρειες, τις τοπικές αρχές. Όχι. Εμείς, εάν υπαρχει σοβαρή περίπτωση, η Ευρώπη είναι στο πλευρό τους. Με οικονομικούς πόρους, με τεχνικό εξοπλισμό, με τεχνογνωσία για να βοηθήσει να απαλληλθούν οι συνέπειες των καταστροφών ή ακόμη και οι συνέπειες των καταστροφών που έχουν προκαλέσει τα άτομα, ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις όσο ταχύτερα γίνεται. Ευχαριστώ. Ο κύριος ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, το θέμα που μας απασχολεί είναι πολύ σημαντικό. Σε κάποιες περιπτώσεις ε, το κράτος μέλος, ένα κράτος μέλος μόνο του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Για παράδειγμα, ο πυρηνικός σταθμός του Αστράβο στη Λευκορωσία. Ξέρουμε ότι η κατασκευή αυτού του πυρηνικού σταθμού έγινε κατά παράβαση των διεθνών προτύπων ε, για το ζήτημα αυτό. Τούτο γίνεται 20 χιλιόμετρα από τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι ε, τεράστιος δυνάμει κίνδυνος. Ζητώ λοιπόν από την Επιτροπή να κάνει ό,τι μπορεί για να υποχρεώσει την Λευκορωσία να σεβαστεί του, τις διεθνείς δεσμεύσεις της και, τις διεθνείς, ε, και τα διεθνή πρότυπα προβλέπει η Επιτροπή να κάνει κάτι τέτοιο, να εξασφαλίσει τους τυχόν, τυχόν κινδύνους από μια καταστροφή. Μετά από πολλές διαπραγματεύσεις φτάνουμε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας γιατί το 2017 και 2018 είχαμε να αντιμετωπίσουμε πυρκαγιές και αποψήλωση των δασών. Ε, θα πρέπει να είναι σε εφελούσια βάση, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συντονίζει τις προσπάθειες όταν μία χώρα ζητά αρρωγή. Αυτό θα γίνει για να μπορέσουμε να ε, διαχειριστούμε καλύτερα και τα μέσα πολιτικής προστασίας. Το RESC-EU, αυτό το αποθεματικό, θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν επαρκή σπόρους και έτσι τα ενδιαφερόμενα κράτη θα έχουν τη δυνατότητα και χρήσης αεροσκαφών για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές. Αυτό αφορά και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ωραία. Αυτή ήταν η τελευταία παρέμβαση. Ο κύριος Στυλιανίδης έχει το λόγο για να απαντήσει και μετά η κυρία Γκαρντίνη. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, όταν πριν από δύο χρόνια ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια. Ειλικρινά υπήρχε μεγάλη προθυμία από πολλά από τα κράτη-μέλη. Και λοιπόν ήξερα ότι είναι πιο σημαντικό να αυξήσουμε το δυναμικό μας. Καθώς και τους πόρους για την προσπάθεια αυτή. Καθώς και το ότι να έχουμε ένα καλύτερο πλαίσιο για την αντιμετώπιση των καταστροφών και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά για μένα και όπως καταλαβαίνω και για σας, το πιο σημαντικό είναι αυτά που επέτυχε συγκεκριμένα το εξής που επέτυχε το Rescue Ενισχύουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Την κάνουμε πιο αποτελεσματική και πιο απτή. Πολύ πιο κοντά στους συμπολίτες μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και ιδιαίτερα στην παρούσα συγκυρία. Τώρα που το κοινό ευρωπαϊκή μας ε, εγχείρημα αμφισβητείται από πολλούς, δυστυχώς. Και ιδιαίτερα επειδή επίκυνται οι πολύ σημαντικέ ευρωεκλογέ. Αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να δώσουμε αποτελέσματα επί των υποσχέσεών μας να κατασκευάσουμε, να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη που προστατεύει, που σώζει ζωές. Είναι ένα μεγάλο επίτευγμα και σας ευχαριστώ και πάλι γι' αυτό. Αλλά μια συμβουλή να σας δώσω. Γιατί συνέλεξα πολύ εμπειρία μέσα από αυτή την κοινή προσπάθεια. Είναι ένα μεγάλο βήμα, αλλά ένα πρώτο μεγάλο βήμα. Πρέπει να συνεχίσουμε για να αναβαθμίσουμε το μηχανισμό αυτό και σε άλλους τομείς. Ιδιαίτερα στον ιατρικό. Αυτό θα είναι ένα επόμενο ορόσημο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Στυλιανίδη. Η κύρια Γκαντίνη, συγγείται, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Άκουσα με πολύ χαρά τις παρεμβάσεις όλων των συναδέλφων και την επιβεβαίωση μιας ενότητας θέσεων και διάθεση συνεργασίας από όλες τις πολιτικές ομάδες, όλους τους βουλευτές, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Σκεφτόμουν και το δρόμο που διανύσαμε από την προηγούμενη θητεία όταν μπήκε η έννοια της πρόληψης μέχρι σήμερα που είναι αναπόσπαστο για να μην πω προτεραιότητα κομμάτι προτεραιότητα στην πολιτική προστασία. Ευχαριστώ τον Επίτροπο που θύμισε τις δυσκολίες να πείσουμε κάποια κράτη-μέλη. Υπάρχει και μία πολιτισμική σεμνότητα να αποδεχθούμε την ανάγκη να ζητήσουμε βοήθεια. Θυμάμαι το δίδαγμα που μάθαμε όταν η Ιαπωνία βρέθηκε μπροστά στην καταστροφή της Φουκουσίμα. Η χώρα που θεωρούσαμε η πιο προπαρασκευασμένη στον κόσμο δεν ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτή την τεράστια καταστροφή. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η σεμνότητα. Η Ευρώπη που προστατεύει που παρακολουθεί είναι μια πραγματικότητα ένα και εντονότερη και χάρη στην προσπάθεια του Επιτρόπου και την δουλειά του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου έχουμε ένα εργαλείο που καθιστά την Ευρώπη ασφαλέστερη. Χαίρομαι που υπήρξε η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε και αυτή τη μεταβατική περίοδο που θα μας επιτρέψει να είμαστε έτοιμοι πριν το επόμενο καλοκαίρι γιατί είδαμε ότι οι μεγαλύτερες καταστροφές αυτές που καταγράφουν το μεγαλύτερο αριθμό απολειών ανθρώπινων ζώων γίνονται πραγματικά το καλοκαίρι με τις δασοπυρκαγιές. Ευχαριστώ επίσης ε, και ξανά όλους σας και αφού αφιέρωσα στον Ζαμπερλέιτ αυτή τη μέρα θέλω να σκεφτώ τις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων που σε όλη την Ευρώπη δουλεύουν για την ασφάλεια όλων μας. Στην πολιτική προστασία, στην πυροσβεστική, στους πάμπολους εθελοντές που σε πολλές χώρες δουλεύουν για μας. Η πολιτική προστασία έχει πολλές μορφές και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο δεν μπορέσαμε να δώσουμε τον ορισμό της πολιτικής προστασίας στην προηγούμενη θητεία. Η ενότητα ωστόσο προθέσεων και αισθημάτων είναι ένα σημαντικό τούβλο για να χτίσουμε την Ευρώπη που αγαπάμε. Μια Ευρώπη που προστατεύει, που έχει μεγαλύτερη λεγγύη και, προσ... βοηθά τους πολίτες σας. Τους πολίτες. Ευχαριστώ όλους για την δουλειά σας. Ευχαριστούμε κύριε Γκαρντίνη. Ολοκληρώνεται η συζήτηση. Συγχαρητήρια σε όλους όσοι ασχολήθηκαν με το φάκελο αυτό και στην εισηγήτρια. Προχωρούμε στην εξέταση της έκθεσης Γκούτελαντ για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Η κυρία Γκούτελαντ δεν είναι εδώ σήμερα. Θα ακούσουμε στη θέση της την κυρία Ντάλι. Μίριαμ, παρακαλώ.